του κανονισμού οι εντολές του κυρίου Αγκουράκη, Στανέλης και Σαραδάκο ελέγχθησαν και προτείνεται ομόφωνα να κηρυχθούν έγκυρες αυτές, οι διορισμοί. Μάλιστα, αφού δεν υπάρχουν ενστάσεις, οι εντολές αυτές επιβεβαιώνονται. Ο κύριος Τσαλίσκι για τις σχέσεις